τις χώρες ε, της Ευρωμεσογειακής Ζώνης, ο κύριος Ντεχούχτ έχει το λόγο. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η νότια γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει διέλθει σημαντικές αλλαγές μετά από το 2011. Μέσα στο αυτό το πλαίσιο, το εμπόριο και οι επενδύσεις <clears throat> πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο ως παράγοντες σταθερότητας στις σχέσεις μας με τις χώρες της νότιας όχθης Μεσογείου. Εστιάζουμε αυτή τη στιγμή σε τρεις κέριους στόχους για την νότια όχθη της Μεσογείου. Ο πρώτος στόχος είναι η εμβάθυνση των εμπορικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους εταίρους μας από την νότια όχθη της Μεσογείου επί τη βάση μιας διαφοροποιημένης προσέγγισης. Το Δεκέμβριο του 2011 ενέκρινε το Συμβούλιο κατευθύνσεις για ιδιαίτερες ε, ρυθμίσεις για την, την Ισία, το Μαρόκο, την Ιορδανία και την Αίγυπτο. Οι συμφωνίες αυτές έχουν σαν στόχο την προοδευτική ενσωμάτωση των οικονομιών αυτής της ζώνης στον χώρο εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι ρυθμίσεις θα καλύψουν τομεί <clears throat> ρυθμίσεως κοινού ε, συμφέροντος όπως είναι η διευκόλυνση του εμπορίου, η υγειονομικά και φυτο υγειονομικα μέτρα, δημόσιες προμήθειες καθώς και πολιτική ανταγωνισμού. Θα απελαμβάνω επίση την προστασία του, των επενδύσεων και τη φιλελευθερωποίηση της εμπορίας αγαθών και υπηρεσιών και της ελευθερίας εγκατάστασης. Οι διαπραγματεύσεις περατώθηκαν με το Μαρόκο το Μάρτιο του το 2013 και συνεχίζουν η πρόοδος των ε, διαπραγματεύσεων είναι μεγάλη με την Ιορδανία και με την Τινησία μπορούν να ξεκινήσουν το ταχύτερο δυνατόν να τελειώσει η διαδικασία προπαρασκευής. Η πρώτη προτεραιότητα για τις χώρες αυτές όπως είναι χώρες όπως η Λιβύα, ο Λίβανος, η Αλγερία είναι να μπορέσουν να συμμετάσχουν και αυτές στο πλαίσιο αυτοσταθεροποίησης. Πρέπει επίσης όμως να βρούμε το καλύτερο πλαίσιο για τη σχέση μας με τη Λιβύη το ταχύτερο δυνατό. Επίσης ένα δεύτερο στοιχείο είναι να υποστηρίξουμε το ενδοπεριφερειακό εμπόριο μεταξύ χωρών της νότιας όχθης Μεσογείου γιατί το ενδοπεριφερειακό εμπόριο είναι χαμηλότερο από ό,τι σε, σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου. Ένα τέτοιο πιο ολοκληρωμένο εμπόριο θα ήταν μεγάλο πλέον πλεονέκτημα. Πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειες για να ενισχυθεί η συμφωνία μεταξύ Αιγύπτου, Ιορδανίας, Μαρόκου και την Ισίας και να ε, επεκταθούν σε άλλους τομείς όπως το εμπόριο υπηρεσιών, οι επενδύσεις και οι δημόσιες προμήθειες. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσουμε και χρηματοδοτική ε, βοήθεια καθώς και παροχή τεχνογνωσίας. Η αναθεώρηση των ε, κανόνων ε, προέλευσης θα πρέπει να επιταχυνθεί. Αυτό δεν είναι εύκολο καθήκον γιατί υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των εταίρων που συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή. Τρίτο στοιχείο είναι η ευρωμεσογειακή εμπορική εταιρική σχέση η οποία θα πρέπει να αναζωογονηθεί στην επόμενη Υπουργική Σύνοδο στις 30 Σεπτεμβρίου της Ευρωμεσογειακής Ζώνης. μια πολύ σημαντική συνάντηση και θα είναι η πρώτη μετά από τέσσερα χρόνια. Κύριε Πρόεδρε, έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Κομισιόν κάνει ό,τι περνάει από το χέρι τη για να διατηρηθούν οι σχέσεις εμπορίου με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου, ε, σε επικαιροποιημένο επίπεδο και να διατηρήσει την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή αυτή. Βασιζόμαστε στην συμμετοχή του Κοινοβουλίου για να πετύχουμε αυτό το κοινό στόχο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Δεχούχτ. Ακολουθούν οι ομιλητές από τα πολιτικά κόμματα. Πρώτη η κυρία Γκάμπριελ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας, για την κατάσταση των πραγμάτων στο εμπόριο με τις χώρες Euromed. Η κατάσταση λοιπόν δείχνει ότι το εμπόριο ανάμεσα στις χώρες μας και στις χώρες του Νότου της Μεσογείου έχει πρόπτικες, αλλά ο δρόμος είναι μακρύς και η εταιρική σχέση δεν θα πρέπει να παραμείνει ασύμετρη. Να υπογραμμίσω εδώ τρία στοιχεία. Πρώτον, είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε τις προσπάθειες που έχουμε κάνει στα πλαίσια της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών. Η κατάργηση των μη δασμολογικών και τεχνικών επιβαρύνσεων θα πρέπει να γίνει με την εμπλοκή και τη συμμετοχή την πλήρη και ισότιμη των χωρών εταίρων. Η συνεργατική αυτή σχέση με τον νότο της Μεσογείου θα πρέπει να βασίζεται σε μια δυναμική ολοκλήρωση. Σήμερα οι ανταλλαγές ανάμεσα στις χώρες του νότου είναι όμως πολύ χαμηλές. Πρέπει να ενισχυθούν επίσης οι εμπορικές συναλλαγές. Έχει σημασία να παραμείνουμε πραγματιστές και να συνεργαστούμε με αυτούς οι οποίοι έχουν δυνατότητες. Σαν παράδειγμα η πολιτική έκδοση θεωρήσεων πρέπει να διευκολύνει τις διαδικασίες για τον επιχειρηματικό κόσμο όπως ακριβώς με τη συμφωνία που υπογράψαμε με το Μαρόκο το 2013, τον μήνα Ιούνιο να διευκολύνουμε την ε, διαδικτύωση των επιχειρήσεων των δύο πλευρών της Μεσογειακής Λεκάνης μέσω διμερών εμπορικών επι, ε, ε, επιμελητηρίων. Και τρίτον, να εμβαθύνουμε τις εμπορικές σχέσεις, όχι όμως σαν αυτό σκοπό. Το εμπόριο δεν είναι η μοναδική κλίδα ανάπτυξης. Είναι όμως κάτι που θα διευκολύνει στις χώρες αυτές να ενταχθούν πλήρως σε μια ανοιχτή οικονομία θα πρέπει εμείς να φροντίσουμε έτσι ώστε η ανάπτυξη των οικονομικών συναλλαγών να ενισχύσει τις κρατικές και διοικητικές δομές των χωρών αυτό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε την αστάθεια, την κοινωνική και οικονομική της περιοχής. Ναι στο εμπόριο, στην υπηρεσία όμως ειρήνης. Σε ευχαριστώ κυρία Γκάμπριελ. Ακολουθεί κυρία Αρένα. Ευχαριστώ κύριε Ντεχούχτ στην παρέμβασή σας δεν αναφερθήκατε στην εταιρική σχέση μεταξύ Ευρώπη και Ισραήλ. Μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσω να υπενθυμίσω ορισμένε αρχέ τη εμπορική μα σχέση για το Ισραήλ, με το Ισραήλ. Καταρχήν, το θέμα τη κατοχή των εδαφών τη ε, δυτική όχθη. Έχουμε εμπορικά εργαλεία τα οποία μα δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε δύο πράγματα. Καταρχήν να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη τα οποία ήδη έχουν πάρει τα απαραίτητα μέτρα για τα προϊόντα τα οποία προέρχονται από τα κατεχόμενα εδάφη τη δυτική όχθη, να μπορέσουν να εξασφαλίσουν ότι υπάρχει σωστή ετικετοθεσία για αυτά τα προϊόντα. Γίνεται με θελοντικό τρόπο. Αυτό έχει γίνει και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Βέλιο. Θέλουμε όμω και σε επίπεδο Ευρώπη να μπορέσουμε να εργοποιήσουμε μέτρα τα οποία είναι δεσμευτικού χαρακτήρα για τη σωστή ετικετοθεσία για τα προϊόντα αυτά τα οποία προέρχονται από τα κατεχόμενα εδάφη τα οποία είναι παράνομα ε, προϊόντα για το Ισραήλ. Αυτό θα επιτρέψει τον Ευρωπαίο καταναλωτή να κάνει τις σωστές επιλογές σε σχέση με την κατανάλωσή του και να αλλάξει τις ε, συνήθειες του καταναλωτικό επίπεδο και να μπορέσει να ασκήσει πίεση για το τέλος αυτής της αδίκης κατάστασης που υπάρχει. Επίσης, ε, επειδή αναφερθήκατε για το Μαρόκο και την Ισία, είναι απαραίτητο και για τις χώρες αυτές να υπενθυμίσουμε ορισμένες αρχές. Καταρχήν, ότι είναι χώρες που είναι σε δημοκρατική μετάβαση, αναφέρομαι περισσότερο στην Ισία, είναι απαραίτητο να μπορέσει να συμμετάσχει και η κοινωνία των πολιτών σε σχέση με τις συμφωνίες αυτής ελευθέρου εμπορίου, να έχουμε κοινωνικές ρήτρες και, και ρήτρες προστασίας του περιβάλλοντος που να είναι και μέσα στα πλαίσια αυτών των εμπορικών συμφωνιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αρένα. Δέχεστε ένα ερώτημα από την κυρία Μορβάη. Δέχεστε ερώτημα από την κυρία Μορβάη. Παρακαλώ κυρία Μορβάη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω ένα ερώτημα για την κυρία Αρένα θα συμφωνούσε μαζί μου ότι πριν από μισή ώρα μιλούσαμε για τη Ρωσία εδώ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποφασίσει ότι η Ρωσία έχει διαπράξει μια εισβολή σε μια άλλη χώρα, μια επίθεση και γι' αυτό θα έπρεπε να εφαρμοστούν κυρώσεις εναντίον της χώρας αυτής. Συμφωνείτε λοιπόν με αυτά τα οποία έλεγχαν ότι είναι σημαντικό να εκφράσετε λοιπόν αυτή την άποψη. Δεν πρέπει να έχουμε δύο μέτρα και δύο, ε, δύο σταθμά. 30 δευτερόλεπτα έχετε μονάχα κύριε Μορβά για το ερώτημά σας, όχι παραπάνω λέει ο πρόεδρος. Μικρόφωνο παρακαλώ. Εγώ μίλησα για την ανιχνευσιμότητα των προϊόντων αυτό επιτρέπει να γίνονται οι επιλογές ανάμεσα στα διάφορα προϊόντα. Αν δεν είναι τέτοιου είδους, ε, ε, δεν υπάρχουν τέτοιου είδους ετικέτες, ε, τότε αυτό θα ήταν λάθος. Εγώ δεν θέλω να απαγορευτούν όλα τα προϊόντα των Ισραηλινών ή των Παλαιστινίων, θέλω να γνωρίζω από πού προέρχονται όμως. Σας ευχαριστώ. Ακολουθεί ο Μαριάς. Ένα λεπτό. Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις μεσογειακές χώρες πρέπει να στηρίζονται στις αρχές του αμοιβαίου ωφέλους και να μην είναι ετεροβαρής. η δημιουργία μιας ελεύθερης οικονομικής ευρωμεσογειακής ζώνης πρέπει να έχει ως στόχο να μην δημιουργεί προβλήματα σε χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα όπως είναι οι χώρες του νότου χώρες που πλήττονται από την μερκελική λιτότητα από τα μνημόνια και αυτό ισχύει και για την ελλάδα και την ιταλία. πολύ δε περισσότερο τώρα που όπως είδαμε η αγροτική οικονομία της ελλάδας και των άλλων χωρών του νότου πλήττονται από το ρωσικό εμπάργκο. επίσης ορισμένες χώρες της μεσογείου δεν πρέπει να έχουν μια πολιτική la carte. αυτό ισχύει για την τουρκία η οποία ενώ έχει εισβάλει στην κύπρο ενώ έχει καταλάβει ένα μεγάλο μέρος του νησιού εν δεν αναγνωρίζει την κυπριακή δημοκρατία και παρά τα αυτά απαιτεί τα προϊόντα της να κυκλοφορούν ελεύθερα και χωρίς εμπόδια στην ευρωπαϊκή ένωση. πρέπει επίσης κύριε πρόεδρε να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα των παράνομων μεταναστευτικών σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το εμπόριο είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της ε- εξωτερικής μας πολιτικής και θα πρέπει να ενσωματώνεται ακόμα περισσότερο σε αυτή την πολιτική. Φάνηκε η σημασία του εμπορίου από την απάντηση στη Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας. ήτανε και ένα, ένας τρόπος αφύπνισης για αυτούς οι οποίοι αγνοούσαν τη σημασία του εμπορίου. Εμείς έχουμε λοιπόν να κερδίσουμε πολλά από το να διευρύνουμε τις, συμφω... τις συμφωνίες που έχουμε στην Ευρωμεσογειακή ζώνη. Μερικά χρόνια μετά από τη στιγμή που πολλοί εξεγέρθηκαν στις χώρες αυτές και ζήτησαν δημοκρατία και ελευθερία, πολλοί από αυτούς νέοι άνθρωποι δεν έχουν επιτευχθεί μεγάλες αλλαγές. Δυστυχώς οι χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα αστάθειας. Παρόλα αυτά εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε φιλόδοξοι στις προσπάθειές μας για το εμπόριο. Πρέπει με τον τρόπο αυτό να δώσουμε νόημα στην έννοια περισσότερα για περισσότερο, περισσότερη πρόσβαση στην αγορά για περισσότερα δικαιώματα ανθρώπινα και δημοκρατία. Θα πρέπει να είμαστε στεναροί στις εξαρτήσεις για το εμπόριο και αυτό αφορά και το Ισραήλ και να δούμε το εμπόριο σαν ένα τρόπο να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη ισότητα, περισσότερα δικαιώματα, να προλάβουμε την ε, άνηση κατανομή του πλούτου και να αντιμετωπίσουμε τη διαφορά και συγχρόνως να ενισχύσουμε και την παιδεία που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπίσει τη μαζική ανεργία των νέων σε αυτές τις περιοχές. Με περισσότερες ευκαιρίες ίσως μπορέσουμε να αποτρέψουμε την ριζοσπαστικοποίηση των ε, νέων εκεί. Και φυσικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα θέματα τη μετανάστευση. Δεν είναι ζήτημα μονάχα καινοτομία και εξαγωγών. Θα πρέπει και ήδη να δούμε ποιο είναι ο αρνητικό αντίκτυπο που έχουν οι εξαγωγικέ επιδόσει στον γεωργικό τομέα για του γεωργού στην Ευρωμεσογειακή περιοχή και τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν. Πρέπει να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο επίση για να εξασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει επικάλυψη των δράσεών μα επιπλέον και να ενισχύσουμε την ε, περιφερειακή ενσωμάτωση που θα βοηθήσει πολύ την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή τη Ευρωμεσογειακή Ζώνη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σάκε. Ακολουθεί για ένα λεπτό ο κύριο Λεγιαρίκ. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, αυτό που ονομάζεται γειτονία με τις χώρες του Νότου της Μεσογείου Κάποιες από τις χώρες αυτές αναζητούν τους δρόμους της δικαιοσύνης ε, και της ελευθερίας. Πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους, όχι να τις ανταγωνιζόμεθα. Είναι απαραίτητο να αλλάξουμε τη στάση μας απέναντι σε αυτές τις χώρες που δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ζώνες διεύρυνσης της οικονομικής μας επιρροής, ούτε χώρες προέλευσης ε, ανθρώπινου δυναμικού χαμηλού κόστους, ούτε επίσης και ζώνες προφυλακτήρες από τα μεταναστευτικά κύματα. Θα πρέπει να σεβαστούμε τις χώρες αυτές, να βοηθήσουμε στις επενδύσεις τους για την αηφόρο ανάπτυξη με κοινωνικές ρήτρες, προσπαθώντας να τις δανειοδοτήσουμε με χαμηλό κόστος και οι πολιτικές συνεργασίες θα πρέπει να συνοδεύονται από σημαντική Πρόοδος πρόοδο στον τομέα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όχι απλά κάποιες προϋποθέσεις για τη βοήθεια σύμφωνα με τα κριτήρια του Δέλτα Νιτάφ. Και η συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ θα πρέπει να διακοπεί μετά από αυτά τα οποία συνέβησαν το τελευταίο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λεγιαρή. Ε, Μπούχνερ για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο γίνεται συνέχεια χειρότερη. Φυσικά ξέρουμε ότι πρέπει να παραμείνουμε σε συνεργασία και σε επαφή με την κυβέρνηση εκεί και να μπορέσουμε να ασκήσουμε στο δυνατόν περισσότερη πίεση για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, η συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την εμπορική συμφωνία είναι κάτι περισσότερο από απλές επαφές ή τεχνικές ε, διευκρινήσεις και συζητήσεις. Αυτό σημαίνει ότι εμείς παραγνωρίζουμε την απώλεια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποστηρίζουμε την κυβέρνηση αυτή και της δίνουμε μια διεθνή αναγνώριση. Για όλους αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πλήττονται από τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα ράπισμα. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω κύριε Επίτροπε κατά πόσο εσείς θα αποφασίσετε να σταματήσετε τις διαπραγματεύσεις μέχρι ότου υπάρξουν πρόοδοι σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στην ε, ε, Αίγυπτο ή τουλάχιστον αναγνωριστεί η δυσκολία αυτής της κατάστασης. Ευχαριστώ για ένα μισή λεπτό η κυρία Μπεγκίν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η συνάντηση των Υπουργών για την Μεσόγειο στις 30 Σεπτεμβρίου θα είναι μια ευκαιρία για να ξανασκεφτούμε τις διάφορες συμφωνίες με τις χώρες της Μεσογείου και να προσπαθήσουμε να δούμε ποια είναι τα συμφέροντα όλων των Ευρωπαίων. Συγγνώμη, δεν έχω γερμανική μετάφραση, λέω Εγώ. Signor Commissario, ho ben noto wait, Excuse me, excuse me, wait, I do not have a... Πρέπει να περιμένετε γιατί υπάρχει πρόβλημα με τη μετάφραση, λέει ο Πρόεδρος. Περιμένετε λίγο. Bitte um entschuldigen, ich habe einen Wackelkontakt. Fangen Sie bitte Ναι, είχα πρόβλημα με την... ήταν ε, κακή επαφή. Τώρα μπορείτε να συνεχίσετε. Η συμφωνία λοιπόν που υπογράψαμε με το Μαρόκο είναι πάρα πολύ ε, γνωστή και πλημμύρισε τις αγορές μας με προϊόντα χαμηλού κόστους ανταγωνιζόμενο χώρες όπως η δική μου και αυτό βοηθά βέβαια κάποιες πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να εξάγουν χωρίς φόρους στο Μαρόκο. Λοιπόν, το θέμα είναι να διαπραγματεύεται η Επιτροπή για την Ευρώπη και όχι για λίγες μεγάλες χώρες και θα πρέπει όλοι οι εταίροι να σέβονται τα διάφορα επίπεδα ε, παραγωγής τα οποία εμείς οι ίδιοι θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει επίσης να δούμε τι γίνεται και με τις συνθήκες εργασίας διότι διαφορετικές συνθήκες εργασίας επικρατούν σε εμά και στις άλλες χώρες της Μεσογείου, κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε κάποια διακανονιστικά πλαίσια που να επιτρέπουν την ασφάλεια των επενδύσεών μας προς τις χώρες αυτές, και να βοηθήσουμε έτσι τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με εγγυήσει, με σωστή ενημέρωση, με δικτύωση, δημιουργώντας τις λεγόμενες διμερείς μορφές εμπορικών επιμελητηρίων με τις χώρες του νότου της Μεσογείου. Τέλος, σας ζητώ να μην ξεχνάμε τον ρόλο του πολιτισμού και των υπηρεσιών στον τομέα του πολιτισμού όπως τον τουρισμό και τα προβλήματα όπως το Εράσμους και τα λοιπά. Είναι απαραίτητα προγράμματα για την ανάπτυξη στο μέλλον της οικονομίας. Από αυτή τη συμφωνία ή θα κερδίσουμε πολλά ή θα χάσουμε πολλά. Από εμά εξαρτάται. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπενιέν. Συγγνώμη για το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισα με την ε, σύνδεση των ακουστικών. Για ένα λεπτό κύριο Σαλιό συνεργασία μεταξύ Ευρώπης, ε, Μεσογείου μάλλον και Ευρωπαϊκών κρατών είναι σημαντικό. Αλλά η κατάργηση στα δική των συνόρων ε, πρώτων οικονομικών και μετά ανθρώπινων μέσω μιας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, όχι. Θέλουμε να υπάρχει ισότιμη ανάπτυξη, αλλά ε, θέλουμε ταυτόχρονα να μειώσουμε τη ροή της μετανάστευσης. Αυτό είναι μια επένδυση για το μέλλον μας, για να στηρίξουμε τις χώρες μας, τους αγρότες, ε, τους ε, εργαζομένους γενικώ. Δεν θα πρέπει με κάθε τίμημα όμως να στηρίξουμε τις νοσογικέ χώρες. Πρέπει και την ασφάλειά μας ε, να την φροντίσουμε ε, βάζοντας όρους, πολιτική σταθερότητα, σεβασμό μειονοτήτων ε, μεταξύ άλλων και κάθε ευρώ που δαπανάται σε αυτές τις χώρες θα πρέπει να φροντίσουμε να χρησιμοποιείται με τοπικό εργοτικό δυναμικό ή αλλιώς από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και να μην χρηματοδοτεί έμεσα την αμερικανική ή την κινέζικη οικονομία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Φίσας Αϊσέλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Οι στόχοι της πολιτικής γειτονίας είναι η δημιουργία ε, μιας ζώνης ευημερίας, σταθερότητας, δημοκρατίας και στόχος είναι και η ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων. Δεν είναι εύκολο το καθήκον, οι πολιτικές, οικονομικές προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι γειτονικές χώρες είναι τεράστιες ε, και η δική μας δέσμευση για να στηρίξουμε τη μετάβαση στις χώρες αυτές προς οι δημοκρατικές κοινότητες πρέπει να είναι σταθεροί και ε, περισσότερο από ποτέ. Υπάρχουν ε, πολλοί λόγοι γι' αυτό, εντονότατες μεταναστευτικές πιέσεις, απειλή για τη σταθερότητα και την ασφάλειά μας, ε, που δημιουργεί αστάθεια, υπάρχει το ενεργειακό ζήτημα που μας κάνει να στρέφουμε το βλέμμα προς τα Μακρέμπ και το οικονομικό δυναμικό που θα είχε η δημιουργία μιας ένωσης μεσογειακής με σταθερές χώρες για την οικονομία μας. Σε αυτή τη διαδικασία αλλαγή το εμπόριο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε ε, τη διαδικασία εμπορικής ένταξης ε, με την άλλη όχθη της Μεσογείου. Και η στις διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες αυτές θα πρέπει οι Κομισιόν να είναι φιλόδοξη στον τομέα τη απελευθέρωση σημαντικού τομεί όπω των υπηρεσιών, των επενδύσεων και των δημόσιων συμβάσεων. Αυτή τη χρονική περίοδο που μεγάλο μέρο των προσπαθειών και των πόρων ε, του εμπορικού θεματολογίου ε, στρέφονται προ άλλε γεωγραφικέ περιοχέ, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να στηρίξουμε την ευρωπαϊκή ε, ολοκλήρωση, την εμπορική μάλλον ολοκλήρωση με τι χώρε τη Ευρωμεσογειακέ. Αυτό πρέπει να είναι προτεραιότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φίσα. Ο κύριος Ταράβελα έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νότιων χωρών της Μεσογείου ξεκίνησε το 1995 με τη διαδικασία τη Βαρκελόνη. Ήταν μια πολιτική, οικονομική και κοινωνική εταιρική σχέση που βασίζεται στην αμοιβαιότητα και την αλληλεγγύη και την συνανάπτυξη. Θέματα τα οποία μα ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Ο σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι απαράγραπτο στοιχείο των συμφωνιών σύνδεση. Η μορφή αυτή τη συμφωνία τονίζει τη σημασία τη οικονομική και εμπορική συνεργασία, αλλά επίση, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, τη συνεργασία σε κοινωνικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Εγώ θα ήθελα μέλο τη Επιτροπή για την ισότητα των φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπενθυμίσω ότι αυτή η συμφωνία, η αυτού του είδου συμφωνία θα πρέπει να είναι ευκαιρία για τη βελτίωση των δικαιωμάτων των γυναικών και ιδίω τη πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση και την απασχόληση και επίση να ενισχύσει τον ρόλο των μέσων ενημέρωση για να τροποποιηθούν και να αλλάξουν νοοτροπίε για την ισότητα ανδρών γυναικών. Θα πρέπει επίση να διευκολύνει τη δημιουργία και την διαχείριση επιχειρήσεων από γυναίκε και την πρόσβαση των γυναικών στα εργαλεία εκπαίδευση. Επαγγελματική και χρηματοδότηση. Επίσης θέλω να χαιρετήσω το θάρρο των γυναικών που ήταν στην πρώτη γραμμή της κοινωνίας των πολιτών και αγωνίστηκαν για τα δικαιώματα των πολιτών και τη δημοκρατία στι Αραβικέ χώρε, δυστυχώ τα αποτελέσματα αυτών των ε, κινητοποιήσεων δείχνουν ότι οι γυναίκες έχουν περιθωριοποιηθεί ακόμα περισσότερο και υφίστανται όλο και περισσότερη βία. όπω και εσεί έχω διαπιστώσει ότι υπάρχουν πολλές πρόοδοι που πρέπει να γίνουν και ελπίζω ότι σέβεστε και εσείς την ιδέα ότι πρέπει να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο ως εταίροι σε αυτές τις εμπορικές συμφωνίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Ταραμπέλα. Ένα ερώτημα από τον κύριο Φεράν, το αποδέχεστε. Κύριε Φερό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ταραμπέλα, υποστηρίζοντας ε, την Αραβική Άνοιξη και τι επαναστάσεις, Μήπως θεωρείτε ότι έχει τεθεί σε κίνδυνο η, η θέση των γυναικών στις χώρες αυτές. Δεν ξέρω αν καταλάβατε πολύ καλά αυτά που είπα κύριε Φερά. Μίλησα για τον κέριο ρόλο των γυναικών στον αγώνα για περισσότερη δημοκρατία, περισσότερα δικαιώματα. Και για τις ίδιες αλλά και για τις χώρες τους. Δυστυχώς είπα, το είπα πολύ σαφώς, ότι δεν μπορούμε παρά να είμαστε απογοητευμένοι από τα αποτελέσματα αυτών των κινητοποιήσεων. Δεν πρέπει σήμερα οι γυναίκε να είναι πιο περιθωρικοποιημένε από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό βλέπουμε και γι' αυτό πρέπει να παίξουμε ένα ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να κάνουμε τα απαραίτητα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση και να μπορέσουν οι γυναίκε να έχουν ένα σημαντικό ρόλο στην οικονομία των χωρών του. Σα ευχαριστώ κύριε Ταραμπέλα. Διαδικασία Catch the Eye και έχει το λόγο κυρία. σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών φοβάμαι ότι η Αραβική Άνοιξη ναι μεν οι γυναίκες έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο δυστυχώς όμως εκ των υστέρων το κίνημα αυτό ε, δεν ακολούθησε μια προοδευτική τακτική. Έχει σημασία να συμφωνήσουμε με τις χώρες αυτές, πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές που βρίσκονται σε μια μεταβατική φάση αλλά θα πρέπει να δούμε μέσω της οικονομίας πώς μπορούμε να επηρεάσουμε πολιτικά. Η διαδικασία της Βαρκελόνης είναι τα θεμέλια της σχέσης μας με τις χώρες αυτές και ένας από τους τομείς συνεργασίας υψηλής σημασίας είναι το περιβάλλον. Είναι προς το συμφέρον όλων να φροντίσουμε την Μεσόγειο θάλασσα, να προστατεύσουμε την Μεσόγειο θάλασσα οι χώρες οι μεμονωμένες μπορούν να κάνουν πολλά μόνες τους, αλλά μεγάλη σημασία έχει η περιφερειακή συνεργασία. Περιμένουμε λοιπόν τη συνάντηση τον μήνα Σεπτέμβριο για να δούμε το τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο τοπικών και περιφερειακών αρχών. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φέλτσερ και Στισέσκου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει και πρέπει να συνεχίσει να το κάνει ένα σημαντικό εταίρο, αλλά θα πρέπει να προσφέρει προοπτικές ολοκλήρωσης σε όλες τις γειτονικές χώρες από την Νότια και Ανατολική Ευρώπη. Προέρχομαι από μια χώρα που υπήρξε κομμουνιστική, ήταν δύσκολη μετάβαση και πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό να παραμένουν ανοιχτά τα σύνορα αν θέλουμε να έχουμε δημοκρατικές χώρες και μιλώ κυρίως για τη νέα γενιά. Μέσω μια συνεχούς συνεργασίας θα μπορέσουμε να φέρουμε τις χώρες αυτές προς τη σωστή κατεύθυνση. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να παρενθούμε τις αρχές μας. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε προσπάθειες γιατί οι πόρτες που έχουν παραμείνει ανοιχτές αντιπροσωπεύουν για τις χώρες αυτές και τη δική τους θέση να σεβαστούν τις δικές μας αρχές. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαδικασία αυτή ε, στα, στα κράτη αυτά. Γιατί αυτό θα οδηγήσει στην ε, ε, σύμπηξη καλύτερων σχέσεων μεταξύ των χωρών αυτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης έχουν πολλά να προσφέρουν σε εμπειρία. Κύριος Γιακοβίτσης έχει το λόγο τώρα. Η πρωτοβουλία αυτή είναι πολύ σημαντική για το νότο της Μεσογείου. Είχα τη δυνατότητα άλλωστε να εκπροσωπήσω την Ευρώπη ε, σε τέτοιου είδους φόρα και κατανοώ τις ανάγκες που έχουν οι φίλοι στη νότια πλευρά της λεκάνης της Μεσογείου. Υποστηρίζω λοιπόν τις διαπραγματεύσεις αλλά να μην ξεχνάμε ότι πρέπει να προσπιστούμε και τα δικά μας συμφέροντα και όχι μόνο ε, εθνικά συμφέροντα αλλά τα συμφέροντα σε επίπεδο αρχών όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα τα οποία υπάρχουν και πρέπει να τα συζητήσουμε αναφέρομαι στο ελαιόλαδο όταν μιλάμε για την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα. Γνωρίζω ότι εισάγουμε πάρα πολύ ε, λάδι, ελαιόλαδο από την ε, ε, Βόρεια Αφρική το οποίο αναμειγνύεται με ευρωπαϊκό ελαιόλαδο και πωλείται ως αμυγός ευρωπαϊκό. Λοιπόν, πρέπει να διορθωθούν αυτά τα πράγματα και να γνωρίσουμε τη χώρα προέλευσης των προϊόντων. Ευχαριστώ. Ο κ. Βίγκας έχει το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο. Μικρόφωνο παρακαλώ. Υποστηρίζουμε τη διαφοροποίηση των σχέσεων μας σε εμπορικό επίπεδο. Αυτό το οποίο ζητάμε είναι να μην είναι μονάχα τα κριτήρια τα οποία ισχύουν μονάχα οικονομικά, δεν είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να μόνα τους να διέπουν αυτές τις σχέσεις. Όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την εξάλληψη των δασμών κτλ. Όλα αυτά βέβαια θα δημιουργήσουν τεράστιες δυσκολίες σε αυτές τις οικονομίες. Όπως ξέρουμε πολύ καλά, έχουμε οδυνηρή εμπειρία στην ε, Πορτογαλία. Θα πρέπει να έχουμε κοινωνικά κριτήρια, κριτήρια που να βασίζονται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο σεβασμό τη κυριαρχικότητα κάθε χώρας και να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε μια λογική συμπληρωματική που θα οδηγήσει σε αμοιβαία ε, ωφέλη για όλε αυτέ τι χώρες. Και επίσης ε, συμφωνώ με αυτό το οποίο ελέγχθη για το Ισραήλ. Είναι ένα παράδειγμα μιας ε, σχέσης όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να παρακάψουμε αυτά τα θέματα, αλλά πιστεύουμε ότι μία από τις λύσεις που μπορούν να δοθούν είναι ένα αποτελεσματικό εμπάργκο. Ένα μονάχα ε, ερώτημα. Σας ευχαριστώ κύριε Βιέγκας, λέει ο πρόεδρος, κύριος Φόιτ. Κύριε Φόιτ. Έχουμε τα θέματα που αναφέρθηκαν για τις βασικές αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρώπη και γι' αυτό θα ήθελα να ξέρω γιατί η Κομισιόν δεν αντιμετωπίζει το θέμα του Ισραήλ. Είναι πάνω από 2.000 νεκροί στη Γάζα και πολλοί από αυτούς είναι παιδιά. Έχει τουλάχιστον 250 σχολεία βομβαρδίσει το Ισραήλ και μεταξύ αυτών είναι καμιά πενταριά σχολεία των Ηνωμένων Εθνών. Μετά σε αυτή την κατάφορη ε, παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της, των συνθηκών για την προστασία του άμυχου πληθυσμού πρέπει να ε, τεθεί σε πάγο η συμφωνία με το Ισραήλ και να σκεφτούμε αν θα πρέπει και να εφαρμόσουμε και εμείς κυρώσεις κατά του Ισραήλ και επίσης να ε, φέρουμε το θέμα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Τελείωσε η διαδικασία του Catch the και κλείνει τη συζήτηση ο Επίτροπος Ντεχούχτ. Merci beaucoup, euh, Monsieur Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ας προσπαθήσω να απαντήσω κάποιες από τις ερωτήσεις οι οποίες τέθηκαν και κάποιες από αυτές τέθηκαν και επανειλημμένα. Για την Αίγυπτο πρώτα. και κάποιοι πιστεύουν ότι δεν θα πρέπει να διαπραγματευτούμε ε, την εμπορική συμφωνία λόγω ακριβώς των προβλημάτων με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς ξεκινήσαμε διαπραγματεύσεις ε, το 2011 αλλά η έναρξη πραγματικά των διαπραγματεύσεων εξαρτάται από την επίτευξη συγκεκριμένων προϋποθέσεων για αλλαγές στη χώρα που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σας ενημερώσει ανάλογα με την πορεία των πραγμάτων. Δεν μπορούμε να διακόψουμε κάτι το οποίο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Τώρα, για άλλες πιθανές εμπορικές συμφωνίες, εμείς έχουμε ξεκινήσει μέσω και εξωτερικών συμβούλων μια αξιολόγηση των δυνατοτήτων των εμπορικών των χωρών αυτών και τις συνέπειές τους σε επίπεδο κοινωνικό και οικονομικό θα υπάρξει ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο για τις επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παράλληλα με τη συνάντηση της 30 Σεπτεμβρίου θα έχω μια διμερή συνάντηση με τον αρμόδιο Αιγύπτιο Υπουργό για το Μαρόκο. Ξέρετε ότι ξεκίνησαν οι, οι της συμφωνίας από το Μάρτιο του 2013. Έχει υπάρξει πρόοδος μέσω των συναντήσεων που έχουν ε, οργανωθεί μέχρι τώρα έτσι ώστε να κλείσουμε μια πλήρη εμπορική συμφωνία το ταχύτερο δυνατόν. Λαμβάνοντας όμως υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα της χώρας αυτής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Μαρόκο έχει ξεκινήσει και κάποιες συνοδευτικές μελέτες σε ορισμένους τομείς για τις διαπραγματεύσεις και έχει συμφωνήσει με την κοινωνία των πολιτών του και τον επιχειρηματικό κόσμο να λάβει υπόψη τα αποτελέσματα των μελετών αυτών κατά τη διάρκεια του επομένου διαπραγματευτικού γύρου. Και γι' αυτό εμείς συζητήσαμε να αναβληθεί ο πέμπτος γύρος. Δεν έχει διακοπεί όμως η διαπραγμάτευση θα συνεχίσουμε τις επαφές κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτής έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Στις 30 Σεπτεμβρίου στα πλαίσια της υπουργικής συνάντησης θα έρθουμε σε επαφή με τους αρμόδιους μαροκινούς υπουργούς. Ελπίζω να μπορέσουμε το ταχύτερο δυνατόν να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία έστω τον επόμενο χρόνο έχει μεγάλη πολιτική σημασία γιατί θα είναι ένα προηγούμενο η συμφωνία αυτή για άλλους εταίρους της περιοχής όπως η Ιορδανία, η Αίγυπτος και η Τινησία. Για το Ισραήλ τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια ξεκάθαρη θέση για, την παράνομη, ε, για τους παρανόμους επικισμούς και για τα προϊόντα τα οποία προέρχονται από τις περιοχές αυτές δεν θα πρέπει να την χάνουν των προτιμησιακών μεταχειρήσεων που προβλέπουν οι συμφωνίες με την χώρα αυτή. Εμείς θα ακολουθήσουμε τις πρακτικές ορισμένων χωρών, αυτό ζητάμε, να διευκρινίζεται η, η σήμανση των προϊόντων αυτών έτσι ώστε να γνωρίζουμε αν τα προϊόντα προέρχονται από τη χώρα του Ισραήλ ή από τους Ισραηλινούς επικισμούς εμείς αναθεωρούμε ε, σταδιακά ε, την ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα της ετικετοθεσίας ιδιαίτερα για τα γεωργικά προϊόντα και θα προτείνουμε σύντομα κάποιες κατευθυντήριες γραμμές στον τομέα αυτό της σήμανσης των προϊόντων έτσι ώστε να υπάρξει μια κοινή λύση. Γενικότερα τώρα έγιναν ορισμένες παρατηρήσεις ε, σχετικά με τη διαδικασία more for more σε όλες αυτές τις εμπορικές συμφωνίες και σε όλες τις διαπραγματευτικές εντολές για διαπραγμάτευση των εμπορικών συμφωνιών θα υπάρξουν ανηλυμένες αμοιβέ υποχρεώσεις στον τομέα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις συμφωνίες αυτές για να προωθήσουμε ε, ισχυρά μέτρα στον τομέα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα προσπαθήσουμε να πείσουμε τις χώρες αυτές σε ε, εθνικό επίπεδο να σεβαστούν τις διαδικασίες του more for more. Ε, υπάρχουν δύο φορές οι λέξεις more όπως είδατε εδώ, δηλαδή περισσότερη βοήθεια, περισσότερες επενδύσεις και περισσότερες πολιτικές αλλαγές. Αυτό σημαίνει αυτή η λογική. Ε, σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να ανοίξουμε και εμείς τις αγορές μας. Αυτό δεν είναι πάντα κάτι το εύκολο που μπορεί να γίνει στα πλαίσια των συμφωνιών αυτών και τα κράτη-μέλη δεν είναι πάρα πολύ ευέλικτα σε σχέση με αυτό. Θα πρέπει επίσης να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε στον τομέα της έκδοσης θεωρήσεων, της χορήγησης θεωρήσεων, που είναι ένας τομέας στον οποίο υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα από πλευρά των χώρων αυτών έτσι ώστε να ανοίξουν και αυτές τις αγορές τους. Πρέπει να αναλάβουν οι χώρες αυτές τις ευθύνε τους, αλλά θα πρέπει και εμείς να κάνουμε το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνε της και να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία από πλευράς μας από ό,τι σήμερα. Ευχαριστώ κύριε Ντεχούχτ. Έχει λήξει η συζήτηση. Στο επόμενο σημείο τώρα έχουμε Κύριε Μορβάη, σας έχω δώσει ήδη μια γραπτή απάντηση στο ερώτημά σας. Εάν δεν ζητάτε το λόγο σε διαδικαστικό